στις 12. Τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης, χωρίς διακοπή, την κατάσταση στη Λευκορωσία. Οπότε, παρακαλώ τον Επίτροπο Πίμπαλξ ως εκπρόσωπο της ΙΑΠ, κυρία Σάστον. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Μεγάλη μου χαρά ε, να συζητήσω σήμερα τη κατάσταση στην Λευκορωσία από πλευράς της υπάτης εκπροσώπου κυρίας Άστον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί όλο και περισσότερο για τη συνεχιζόμενη έλλειψη σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στην ε, Λευκορωσία. Τους τελευταίους μήνες η κατάσταση έχει πάει το κακό στο χειρότερο. Περαιτέρω κατασταλτικά μέτρα και πολιτικέ ε, εναντίον τη κοινωνία των πολιτών και την πολιτική αντιπολίτευση. Έχουμε πολλέ ανησυχίε. Η πρώτη από, από αυτέ είναι ότι θέλουμε αμέσω και χωρί όρου να απελευθερωθούν και να αποκατασταθούν και οι 12 πολιτικοί κρατούμενοι. Η παρουσία πολιτικών κρατουμένων, η ύπαρξη πολιτικών κρατουμένων στην καρδιά τη Ευρώπη είναι έσχος. Επίσης ε, υπάρχουν ε, αναφορές σε βασανιστήρια και απάνθρωπες ηθίκε κράτηση. Καλούμε τι αρχέ τη χώρα να σεβαστούν πλήρω την απαγόρευση των βασανιστήριων και οπωσδήποτε να διερευνήσουν ε, αυτά που έχουν ακουστεί προ αυτήν την κατεύθυνση. Όλε οι πιέσει προ τα μέλη τη αντιπολίτευση και τη κοινωνία των πολιτών πρέπει να σταματήσουν. Και δεν είναι δυνατόν να περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του. Η όλο και πιο δρακόντια νομοθεσία θα περιορίσει περαιτέρω την ελευθερία συνέρχεστε και συνεταιρίζεστε των πολιτών, καθώς και την παροχή στήριξης στην κοινωνία των πολιτών. Όλα αυτά πρέπει να ανατραπούν. Η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που ακόμη εφαρμόζει τη θανατική ποινή. Όπως ήδη είπα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εναντίον της θανατικής ποινής σε όλες τις περιπτώσεις. Σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Της 16 Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τι αρχές της Λευκορωσία να μην υπάρξουν εκτελέσεις του Τσμίτρη Καναβάλοφ και του Λάντισλαβ Καβαλιόφ και να υπάρξει μορατόριο, μορατόριο για τις ε, θανατικές με στόχο την τελική κατάργηση τη θανατικής ποινή. Η πολιτική μας βασίζεται σε αρχές. Δεσμευόμαστε για μια ορατή και ενωμένη υποστήριξη των αρχών μας ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδει ελευθερίε, κράτο δικαίου. Είναι σαφέ ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδρανεί, διαπιστώνοντα εξελίξει σε μια χώρα που είναι γείτονα τριών κρατών μελών. Τα περιοριστικά μέτρα τη Ένωση είναι σημαντικό εργαλείο για να διατηρηθεί η πολιτική πίεση στην Μπελαρούς για να ε, ενισχύσουμε το πολιτικό μας μήνυμα προς την Λευκορωσία. Η Ένωση έχει επανειλημμένα τονίσει ότι όλα αυτά τα μέτρα μπορούν να αναθεωρηθούν ανα πάσα στιγμή. Τον Ιανουάριο το Συμβούλιο διεύρυνε τα κριτήρια για να τιμωρήσουμε όλου όσου είναι υπεύθυνοι για σοβαρέ παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τις, ε, την ε, καταστολή τη κοινωνία των πολιτών και επίση για όλα τα άτομα που ωφελούνται ή υποστηρίζουν το καθεστώ. Όπω είπε και η κυρία Άστον, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών του Φεβρουαρίου, Συνεχίζουμε τις εργασίες μας με στόχο να υπάρξει μια απόφαση στο Συμβούλιο Εξωτερικών της 23 Η Μαρτίου με βάση ένα κατάλογο επιχειρηματικών συμφερόντων που υποστηρίζουν το καθεστώς ή υποφελούνται από αυτό. Καταστήσαμε σαφε ότι οι πολιτικές της Ένωσης δεν ε, στοχεύουν την Λευκορωσία αυτή καθεαυτή, ούτε βέβαια το λαό τη. Η Ένωση διατηρεί την πολιτική κριτικη εμπλοκη μέσω διαλόγου, και μέσω της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε τις διμερείς σχέσεις ανάλογα με την πρόοδο που θα γίνει από τις αρχές όσον αφορά το σεβασμό των αρχών της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Όπως είπε μεταξύ άλλων ε, η κυρία Άστον στην κοινή δήλωσή της με την Υπουργό Εξωτερικών Κλίντον στις 18-12 του η Ένωση παραμένει αποφασισμένη και διατεθειμένη να βοηθήσει την Λευκορωσία να ανταποκριθεί στι υποχρεώσει στον τομέα αυτό. Η εμπλοκή μα με την ε, κοινωνία των πολιτών στη Λευκορωσία, την πολιτική αντιπολίτευση και το κοινό γενικά είναι ζωτικό στοιχείο τη πολιτική μα. Είμαστε διατεθειμένοι ακόμη να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει για διευκόλυνση θεωρήσεων και συμφωνίε επανεισδοχή που θα ενισχύσουν την επαφή μεταξύ ανθρώπων προ όφελο του πληθυσμού τη Λευκορωσία. Δυστυχώ, οι αρχέ τη χώρα μέχρι στιγμή δεν έχουν ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μα για έναρξη διαπραγματεύσεων. Επίση, θα ενισχύσουμε το διάλογό μα με την κοινωνία των πολιτών και την πολιτική αντιπολίτευση μέσω ενό ευρωπαϊκού διαλόγου εξυγχρονισμού με την κοινωνία τη χώρα, για τι αναγκαίε μεταρρυθμίσει, για τον εξυγχρονισμό τη χώρα και για τις σχετικές εξελίξεις, τη σχετική αύξηση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υποστηρίξουμε όσο μπορούμε αυτές τις προσπάθειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θέλουν να αποκτήσουν περισσότερη επαφή με τη Λευκορωσία και να συμμεριστούν την επιτυχή πείρα τους μετάβαση στην ε, δημοκρατία και την οικονομία της αγοράς. Όταν θα είναι όριμες συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να παράσχει στις ε, εταιρείε μας και τα χρηματοπιστωτικά μας ιδρύματα τις αναγκαίες συνθήκες για να υποστηρίξουν την μετατροπή της χώρας και να επενδύσουν στη διαδικασία ιδιωτικοποίηση τη Λευκορωσία. Ο Ευρωπαϊκό Διάλογο θα ξεκινήσει στι Βρυξέλλε στι 29 Τρίτου. Θέλουμε να επιτύχουμε μια ανοιχτή συζήτηση όπου θα συμμετάσχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και η κοινωνία των πολιτών με σημαντική συμμετοχή από τα κράτη-μέλη. Είναι δύσκολη καιρή. Είναι σημαντικό λοιπόν να διατηρούμε κανάλια επικοινωνία και ενημέρωση. Γι' αυτό η Ένωση αναβάθμισε την εκπροσώπησή τη στο Μίνσκ πέρυσι το καλοκαίρι. Κατόπιν ε, του αιτήματο ε, των αρχών τη χώρα αυτή στι 28 Φεβρουαρίου ότι ο επικεφαλή τη ε, αντιπροσωπεία τη Ένωση και ο πρέσβη Πολωνία θα πρέπει να φύγουν από τη χώρα για διαβουλεύσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε μια αποφασιστική ενέργεια αλληλεγγύη να αποσύρει όλου του πρέσβει τη Ένωση για διαβουλεύσει. Οι πρέσβει μα παίζουν ένα ζωτικό ρόλο επιτόπου στη Λευκορωσία. Είναι κανάλια επικοινωνίας και ενημέρωσης και είμαστε πάντα δεσμευμένοι σε μια ενωμένη και συντονισμένη προσέγγιση και του θέματος της επιστροφής τους. Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα που να μας ενθαρρύνει να αλλάξουμε την πολιτική μας έναντι των αρχών στο Μίνσκ. Δεν έχουν απελευθερωθεί πολιτικοί κρατούμενοι, ούτε έχουν αποκατασταθεί. Οι διώξει κατά ηγετών της αντιπολίτευσης από τις εκλογές του 2010 και μετά συνεχίζουν. Οι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχίζονται. Και βεβαίως, περαιτέρω κυρώσει δεν θα βελτιώσουν μάλλον τις διμερείς μα σχέσεις με το Μίνσκ. Λυπηρό αυτό. Αλλά και αναπόφευκτο. Αν θέλουμε να παραμείνουμε πιστοί στι αρχέ μα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ του βουλευτέ για την αποφασιστικότητά του να αντιμετωπίσουν αυτό το δύσκολο θέμα κατά μέτωπο. Το οφείλουμε στο λαό τη Λευκορωσία. Να του δόξουμε, να του δείξουμε την αλληλεγγύη μα μαζί του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και ότι θα έχουν ευρωπαϊκό μέλλον όταν το επιτρέψουν οι συνθήκε. Η υποστήριξη των ε, βουλευτών για την εξελισσόμενη κατάσταση στον Μπελαρού από τι 19 του 10, όταν είχαμε προεδρικέ εκλογέ, ήταν ζωτική σημασία ώστε αυτό το θέμα να παραμείνει ω υψηλή σημασία θέμα στην ημερήσια διάταξή μα. Ζωτικό επίσης για να διατηρήσουμε την πολιτική πίεση επί της χώρας για να αλλάξει η, σημερινή κατασταλτική της πολιτική και να λάβει τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να μπορέσει να βρει τη θέση που της αρμόζει στην Ευρωπαϊκή Συνεργασία. Θα εξετάσουμε το ψήφισμά σας όταν θα το εγκρίνετε αύριο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. Οι εκπρόσωποι των ομάδων τώρα. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για την ε, μακροσκελή, εξαντλητική και πραγματικά πολύ δική και οξυδερκή δήλωση για την ε, Λευκορωσία. Φαίνεται από την έκθεσή σας ε, για τη Λευκορωσία ότι η εσωτερική κατάσταση στη χώρα αυτή δεν έχει βελτιωθεί. Μάλιστα είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ συχνά. Ε, Επανειλημμένως ε, ζητήσαμε την ε, κατάργηση της θανατικής ποινής στη Λευκορωσία. Σήμερα μιλούμε για την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διπλωματικό πόλεμο που κήρυξε η Λευκορωσία πριν από δύο εβδομάδες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί με τον διπλωματικό αυτό πόλεμο χαμένη θα βγει η Λευκορωσία. Ε, ελπίζω να μην ε, βγει κανένα ε, χαμένο και ιδιαίτερα ο λαό τη Λευκορωσία. Γιατί μια τέτοια προοπτική είναι πολύ ζωφερή. Μοναδική συνέπεια ενό τέτοιου διπλωματικού πολέμου θα είναι η ενίσχυση τη δυσάρεση αυτή τη κατάσταση που επικρατεί ούτω ή άλλω στο εσωτερικό τη Λευκορωσία. εξακολουθεί να υπάρχει διαδικασία ε, βελτίωση κατάστασης. Ελπίζω να επανέλθει η Λευκορωσία ε, σε στοιχειώδεις ε, σχέσεις με τις δυτικές χώρες, ε, αλλά γι' αυτό είναι απαραίτητο να αποφυλακίσει τους πολιτικούς κρατευμένους, να σταματήσει την καταστολή κατά της αντιπολίτευσης, να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθεροτυπία και την ελευθερία των δημοσιογράφων. Αυτές είναι οι στοιχειώδεις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι, ήρθε η ώρα για τις αλλαγές, αυτό είναι το μήνυμα προς το ΜΙΣΚ, αρκεί να μην είναι πολύ αργά ήδη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στο ψήφισμά μας, όπως είπε ο κύριος Προτάσεβιτς, ε, φαίνεται ότι το καθεστώς Λευκορωσίας επιλέγει την αυτοαπομόνωση. Δυστυχώς απομονώνει τη Λευκορωσία, αλλά όχι μόνο το κράτος, απομονώνει και το λευκορωσικό λαό. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο, ούτε από εμάς. Αυτό λέμε και στο ψήφισμά μας. Αυτό λέμε και στο ε, αίτημά μας για επίδειξη αλληλεγγύης προς τον λευκορωσικό λαό. Θέλουμε να δείξουμε την αλληλεγγύη μας για να αντιληφθεί ο λευκορωσικός λαός ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε αλληλέγγυοι προς τους λευκορώσους και εκφράζουμε τη βοήθεια και την ελπίδα μας ότι Αντίστοιχα και η Λευκορωσία και ο λαός της Λευκορωσίας και οι λευκορωσικές αρχές θα κάνουν μια χειρονομία προς ε, περισσότερη δημοκρατία, κράτος δικαίου και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η λευκορωσική οικονομία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη φάση. Αν δούμε το έλλειμμα του προϋπολογισμού, το έλλειμμα στο συζύγιο προϊόντων και τις μελλοντικές προοπτικές, βλέπουμε μια ζωφερή εικόνα. Δεν υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης χωρίς μεταρρυθμίσεις και οι μεταρρυθμίσεις είναι αδιανόητες χωρίς προηγούμενη αλλαγή της νοοτροπίας στην κοινωνία χωρίς ένα ε, έναρξη διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, με νέους, με ανεξάρτητες ομάδες, με δημοσιογράφους και με συνδικάτα. Μόνο έτσι μια κοινωνία όποια και αν είναι, είτε στη Λευκορωσία είτε οποιοδήποτε αλλού, μπορεί να είναι σταθερή. Μόνο έτσι και η κοινωνία και η οικονομία μπορούν να συμβαδίσουν και να βελτιωθούν. Αυτό είναι το περιεχόμενο του ψηφίσματός μας. Βέβαια, ε, περιλαμβάνεται φυσικά στο ψήφισμα και το αίτημά μας να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι άσχετα από την πολιτική παράταξη από την οποία προέρχονται. Αυτό είναι το αίτημά μας, αυτό λέει το ψήφισμά μας, που μάλιστα είναι και κοινό ψήφισμα. Δεν είναι δηλαδή μόνο ψήφισμα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, αλλά όλων των Δημοκρατικών Πολιτικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιούλαντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομάδα μου χαιρετίζει την σωστή απόφαση των κρατών μελών να μετακαλέσουν τους πρέσβεις από το Μίνσκ για διαβουλεύσεις μετά τη διπλωματική διαμάχη ανάμεσα στην Ένωση και την Πελαρούς. Η συμπεριφορά του Πρόεδρου Λουκασέγκα και εθνικά και διεθνώ είναι σκανδαλώδη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να τον κολακεύει αυτόν και τα φιλαράκια του, στέλνοντα εκπροσώπους στο Μίνσκ σε επίπεδο πρέσβεων. Ο Λουκασέγκα συνέχεια αγνοεί τις διεθνείς δεσμεύσεις της Μπέλαρους ως, μέλος, μέλους του ΑΣΕ και εγώ δεν θα ήθελα οι διακεκριμένοι πρέσβεις της Ένωσης να παρουσιάζουν τα διαπιστευτήριά τους σε έναν εγκληματία δικτάτορα δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδο στη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Λευκορωσία πριν το καθεστώ αρχίσει οι δημοκρατικέ μεταρρυθμίσει. Μέχρι τότε θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τι προσπάθειέ μα στο να έρθουμε σε επαφή με την ε, κοινωνία των πολιτών και τη δημοκρατική αντιπολίτευση. Επίση, θα ήθελα να ενθαρρύνω τη Διεθνή Ομοσπονδία Ice Hockey να μετακινήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2014 από τη Λευκορωσία κάπου αλλού. Ο Λουκασέγκα δεν αξίζει την τιμή να προεδρεύσει στην ανακτήρια τελετή. Ένας δικτάτορας που δεν καταλαβαίνει τις αρχές της δημοκρατίας, σίγουρα δεν καταλαβαίνει ούτε τις αρχές του αθλητισμού. Την αρχή του ελεύθερου και ε, τίμιου ανταγωνισμού και άμυλα. Σε ευχαριστώ. Κυρία Συνάδελφα. Ο κύριος Βένα Σούλτς. Πρόεδρε Συνάλφου, η Λευκορωσία είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την νοθεία που, με την οποία επανεξελέγει ο κ. Λουκασέγκο αντιμετωπίζει την αντιπολίτευση με βία και τρομοκρατία. Άτομα που το μόνο του αδίκημα είναι ότι έχουν ζητήσει δημοκρατία και να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων, τους βασανίζουν, ψεύτικη η ομολογία, τους κλείνουν στη φυλακή. και θα μπορούσαμε επιπλέον να παγώσουμε τους εξωτερικούς λογαριασμούς των ατόμων που συνδέονται με το καθεστώς αυτό και να στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών. Αλλά πρέπει να δούμε σε τι βαθμό τα μέτρα αυτά θα έχουν επίπτωση. Σε τι βαθμό δηλαδή, για παράδειγμα, ο Υπουργός Εσωτερικών της Μπελαρούς μπορεί να πάει στην ε, διάσκεψη Ιντερπολ στην Λιόν και διάφοροι άλλοι κοντινοί στο δικτάτορα μπορούν να ταξιδεύουν ως μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Θα πρέπει να δούμε γιατί τα επιτρέπουμε αυτά. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ε, στη Μπελαρούς είναι κρατικές. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ε, με 6 δισεκατομμύρια πλεόνασμα στις εμπορικές μας σχέσεις, πλεόνασμα για τη Λευκορωσία προς τη χώρα αυτή, είμαστε από τους κυριότερους υποστηρικτές οικονομικά. Πρέπει λοιπόν τα μέτρα μας να μην θίγουν τα άτομα. Θα πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις κατά συγκεκριμένων μέσα ζώντων και επιχειρήσεων. Για παράδειγμα για τις εξαγωγές λιπασμάτων, χάλιβα, για να μπεκοτάρουμε ή να μετακινήσουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ice Hockey δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο θα ήταν ε, ικανοποιητικό αυτό το γεγονός αλλά νομίζω ότι θα είχε αρνητική επίπτωση για τον πληθυσμό και για την εικόνα του δικτάτορα, όπως είδαμε και το 80 με την Μόσχα. Διότι αν θέλαμε να είμαστε συνεπείς, τότε δεν θα έπρεπε να δεχτούμε και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Ευχαριστώ τώρα. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Μιγκάλσκι. Σας ευχαριστώ. Το ψήφισμα για τη Λευκορωσία είναι καλό ψήφισμα γιατί επισημαίνουμε και παραλαμβάνουμε κάτι που ανέκαθεν τονίζαμε. Τη διατήρηση των οικονομικών κυρώσεων, το αίτημα για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, την εξασφάλιση των στοιχειωδών προϋποθέσεων για πολιτική συνεργασία δηλαδή ελευθερία στην κοινωνία των πολιτών, αποφυλάκηση των πολιτικών κρατουμένων, επαναλαμβάνω, ε, αναφέρθηκε το επίθετο Μπανταρεύκη και Σιβιόσουφ. Έχω προσωπικές επαφές ε, με τους ε, δύο κρατουμένους αυτούς και το πιο σημαντικό είναι ότι καλό είναι να ε, επισημαίνουμε από καιρού καιρών ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε στη ε, Λευκορωσία τα ελεύθερα μέσα μαζική ενημέρωση. Μόνο με ελευθεροτυπία θα αλλάξει η κατάσταση στη Λευκορωσία και με ελεύθερε εκλογέ να μπορέσουν αργά ή γρήγορα να εκφράσουν την ελεύθερη του ε, πολιτική βούληση οι πολίτε τη Λευκορωσία. Αυτό είναι κάτι καινούριο και θα πρέπει να του δώσουμε την απαραίτητη προσοχή. Σε αντίθεση με κάποιου προλαλήσαντε, εγώ θεωρώ ότι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ε, αυτό το αίτημα για αλλαγή της ε, διοργάνωσης ε, και μεταφορά του παγκόσμιου προσταθλήματος και επιπάγου από τη Λευκορωσία κάπου αλλού. Είναι αδύνατον να έχουμε ένα τέτοιο σημαντικό αθλητικό γεγονός σε μια χώρα που εφαρμόζει βασανιστήρια κατά των πολιτικών κρατουμένων, κατά των μελών της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του ψηφίσματός μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάριν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Έχω τέσσερα παιδιά στην οικογένειά μου. Όταν ένα από τα παιδιά μου έρχεται, τα άλλα φεύγουν, ε, γιατί κάπου έχουν να πάνε. Bad στην περίπτωση της ε, Λευκορωσίας, τα πράγματα δεν είναι, είναι, είναι κάπως έτσι, είναι σαν να μιλάς με μικρά παιδιά. Ε, τελικά είναι σαν να πιέζουμε την, ε, την Λευκορωσία να πάει κάπου αλλού. Αυτό το κάπου αλλού είναι η Ρωσία. Τα τελευταία χρόνια το εύρος της δημοκρατίας έχει συσταλεί, έχει συρρυκνωθεί αντί να διευρυνθεί. Αντί να φέρουμε την Λευκορωσία κοντύτερα στην Ευρώπη, την απομακρύναμε. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να κινηθούμε με σοφροσύνη και προσοχή. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το καρότο και το ραβδί. Το καρότο θα μπορούσε ας πούμε να είναι η αύξηση της οικονομικής μας συνεργασίας με την Λευκορωσία αντί να την μειώσουμε, να την αυξήσουμε λοιπόν έτσι ώστε να αυξηθεί ε, η ευμάρεια Ε, όπως και στην ε, Βόρεια Αφρική, ε, διαπιστώνουμε και στη Λευκορωσία ότι η μεσαία τάξη προσδοκά την δημοκρατία. Και βεβαίως, από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να απαιτήσουμε σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κύριε Σβήγενον. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Ο λόγος για τον οποίο έχουμε τη συζήτηση αυτή σήμερα είναι γιατί οι κυρώσεις κατά του καθεστώτος Λουκασέγκα παρατάθηκαν άλλη μια φορά και αυτό οδήγησε σε μια διπλωματική διαμάχη μεταξύ της Ένωσης και της ε, Λευκορωσίας. Χαίρομαι πολύ που εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αποστήλαμε ένα σαφές μήνυμα προς το καθεστώς ε, Λουκασέγκα ότι είναι απαράδεκτο να ασκούνται πιέσει σε μεμονωμένα κράτη της Ένωσης. Διότι η Ένωση λειτουργεί συνολικά. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τη χώρα αυτή, την πορεία προς τη δημοκρατία. Τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, και το να μην υπάρξουν εκ νέου λήψεις. Τι μπορούμε να κάνουμε ούτω ώστε μετά τις εκλογές, ε, συγγνώμη, οι επόμενε εκλογές να είναι κάπως ε, λιγότερο ε, άδικες, με λιγότερη νοθεία, πιο δημοκρατικές. Νομίζω πως δεν είμαστε αρκετά δημιουργικοί. Διότι είτε παρατείνουμε κάθε φορά τις κυρώσεις είτε κάνουμε στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις είτε προτείνουμε τέτοιες στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις που δεν θα θίξουν τον πληθυσμό της ε, χώρας αυτής. Δυστυχώς όμως αναφερθήκαμε και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα χόκι επιπάγου. Δεν νομίζω ότι μπορεί τώρα να πάει αλλού τώρα πια. Αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε να οδεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση και ελπίζω ειλικρινά ότι κάτι θα επιτύχουμε διότι οπωσδήποτε πρέπει να ε, βοηθήσουμε περισσότερο τη χώρα αυτή. Ο κύριος Γκουτμάνης, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε το ψήφισμα αυτό, κυρίως δε το τμήμα των κυρώσεων κατά αυτών που φέρουν την ευθύνη για την καταστολή, που, ε, καταστολή πολιτικών αντιπάλων τους στην ε, Λευκορωσία καθώς επίσης ε, και την συρρήκνωση της κοινωνίας των πολιτών. Ε, υπάρχει βέβαια και το σημείο αυτό για το, ε, για το ε, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χοκκί Επιπάγου. Με αυτό δεν συμφωνώ. Πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν τελευταία στιγμή να κάνουμε κάτι τέτοιο. Είναι σημαντικό επίσης να κατανοήσουμε ότι πολλοί θα πάνε στην Λευκορωσία λόγω ακριβώς του πρωταθλήματος χοκκί επιπάγου και θα έχουν τη δυνατότητα ενδεχομένως να έχουν μια ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων ε, και πληροφοριών ε, με τους πολίτες της Λευκορωσίας. Στην ουσία αυτό θέλουμε κι εμείς. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει αυτό το προδάστημα να γίνει τμήμα της λύσης και όχι του προβλήματος. Ευχαριστώ κύριο Σκόβαλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι η ώρα να δούμε ποια ήταν τα τελευταία χρόνια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Λευκορωσίας τι χαρακτηριστικά είχε και πώς την αντιλήφθηκε η, ε, η, η εξουσία στο Μίνσκ. Ε, ψευδεστήσεις, παραπλάνηση, παρεστήσεις, τελείως εσφαλμένη εντύπωση είχε το Μίνσκ και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Θα πρέπει λοιπόν να σταθούμε λίγο και να αναλύσουμε αυτή την πολιτική και να ε, υιοθετήσουμε μια συνεπή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει τα κράτη-μέλη να, ε, να έχουν αντιφατικές πολιτικές, να μιλάμε ε, μεταξύ μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διμερώς να έχουμε εμπορικές επαφές ε, με τη Λευκορωσία. Σήμερα το σημαντικότερο είναι να υποστηρίξουμε την αντιπολίτευση ε, κατά του Λουκασέγκο, γιατί η αντιπολίτευση είναι η πραγματική εταίρη μας. Ο Λουκασέγκο θα πρέπει να ακούσει από εμά ότι αν υπάρξει νέα θέρμανση εντό εισαγωγικών, ε, θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα αν θέλει αναθέρμανση των σχέσεων. Ελευθεροτυπία, ελευθεροτυπία στο ελευθερία στο διαδίκτυο, χωρίς όρους. Αλλιώς ε, ποτέ δεν πρόκειται μόνο στο να αλλάξει την θέση του, ούτε να εφαρμόσει ελεύθερες εκλογές. Και ακόμη και επόμενε εκλογές να γίνουν, πάλι το ίδιο θα γίνει. Κάθε μισό ε, χρόνο θα έχουμε αλλαγή τη πολιτικής και ε, ψευδεστήσει πάλι. Αυτό παίζει, αυτό αυτό το παιχνίδι παίζει ο Γουκασέγκο για να μα ρίξει στάχτη στα μάτια και να συνεχίσει την καταστολή τη ε, αντιπολίτευση. Θα πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική μα. Η κυρία Βάιντερ, η κατάσταση στη Λευκορωσία έχει επιδεινωθεί σοβαρά. Το καθεστώς καταδιώκει και καταστέλει την, τους εκπροσώπους ε, του τύπου και άλλους εκπροσώπους των πολιτών. Μετά από μια εντελώ άδικη δίκη, δύο εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης έχουν καταδικαστεί σε θάνατο, κρατούνται σε κάπου μυστικά Η κυβέρνηση ελπίζει ότι η αντίδρασή μας θα εξαρτηθεί από την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων. Η Λευκορωσία είναι μικρή χώρα. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τις δικές μας προδιαγραφές. Ε, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο στις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Πρέπει να έχουμε πολύ στοχευμένες κυρώσεις για κάποια μέλη του καθεστώτος. Ε, πρέπει να παγώσουμε ε, τα περισσότερα του στοιχεία στις Ευρωπαϊκές Τράπεζες, να τους απορρέσουμε να ταξιδεύουν. Πρέπει να στοχεύσουμε άτομα και εταιρείε που υποστηρίζουν το καθεστώ, αλλά όχι τα άτομα, όχι τι μικρέ επιχειρήσει. Αν σταματήσουμε να συνεργαζόμαστε με τη Λευκορωσία, τότε ο λαό θα την πληρώσει. Οπότε θα στραφούν εναντίον μα, αντί να του κάνουμε συμμάχου μα. δεν θα θεωρήσουν ότι του αντιμετωπίζουμε σωστά. Πρέπει λοιπόν να του υποστηρίξουμε και να υποστηρίξουμε γενικά την κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ο κύριο Παλέτσκι. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, η ανάκληση πρέσβεων ήταν μέτρο που ε, συνηθιζόταν. Αλλά η Λευκορωσία έχει πάντα την επιλογή. Μπορεί να αυτοαπομονωθεί. Είναι ένας κίνδυνος. Οι επικείμενες εκλογές και πάλι δεν θα επιτρέπουν καμία επιλογή. Πώς να ευνοηθεί η σχέση με την Ένωση, μόνο αν απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι και αν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, έστω και σταδιακά βεβαίως. οι σημαντικότεροι εταίροι μας, ε, η Ρωσία και η Ευρωνέστ, πρέπει να πιέσουν και αυτή την Λευκορωσία προς αυτή την κατεύθυνση. Να μην επιδεινώσουμε περαιτέρω τις σχέσεις. Διότι θα υποφέρει ο πληθυσμός αν το κάνουμε αυτό. Οι χώρες της Ένωσης πρέπει να συνεχίσουν να διατηρούν επαφές με την Λευκορωσία, αλλά το μέλλον της Λευκορωσίας θα αποφασιστεί βέβαια εντός της χώρας αυτής οι πολίτες. Πρέπει να είναι πιο ενεργοί στο εγγύς μέλλον. Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης και οι δημοσιογράφοι τον τελευταίο καιρό δεν είχαν καμία δυνατότητα να ταξιδέψουν έξω από τη χώρα. Και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να ισχύει αυτή η καταστολή κατά των δημοσιογράφων. Η Ένωση λοιπόν πρέπει να καταγγείλει το Μίνσκ, διότι η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων είναι μία από τις βασικές ελευθερίες των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Κασμάρεκ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Ήδη στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης συνεχάρει την εκπρόσωπο πολυδιάστων γιατί αυτή τη φορά οι αποφάσεις για τη Λευκορωσία ήταν άμεσες, μονοσήμαντες και απτές. Όλα δείχνουν ότι η αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε εντύπωση και στον πρόεδρο της Λευκορωσίας. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, ίσως τελικά ε, βρήκαμε έναν, μεθο... έναν αποτελεσματικό τρόπο στις δράσεις μας με τη Ρωσία. Ο τρόπος αυτός είναι να εφαρμόζουμε τέτοιες δράσεις που θα πονάν πραγματικά εκεί που ε, θα πονάνε τη Λευκορωσία στα πιο ευαίσθητα σημεία. Ε, ο κύριος και είπε ότι δεν θα πρέπει η Λευκορωσία να διοργανώσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χόκκι Επιπάγου το 2014, γιατί αυτό θα είναι μια ευκαιρία για τον Λουκασέγκο να προβληθεί και να παρουσιάσει τη Λευκορωσία ως κανονική φυσιολογική χώρα στην οποία λαμβάνουν χώρα κανονικέ αθλητικές εκδηλώσει. Αυτό δεν ισχύει. Δεν είναι κανονική φυσιολογική χώρα η Λευκορωσία από τη στιγμή που παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει κράτο δικαίου και δεν μπορεί ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα να εφαρμόζεται σε μια τέτοια χώρα χώρα η οποία στερεί από τους πολίτες τις στοιχειώδεις ελευθερίες και δικαιώματα. Γιατί ε, ε, μια τέτοια διοργάνωση ε, δεν θα φέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα όπως συνέβη με τους Ολυμπιακούς ε, Αγώνες στην Κίνα που δεν είχαν καμία, κανένα αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να ξεσκεπάσουμε αυτή την ψευδεπίφαση της κανονικότητας που προσπαθεί να προβάλλει ο Κουκασάνικο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Μαυρονικόλας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σοσιαλιστική ομάδα τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτή η εταιρική σχέση θα προωθήσει τους δημοκρατικούς θεσμούς, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη μεταρρύθμιση στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα. η ευρωπαϊκή ένωση έχει ως στόχο να επιτύχει πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στη λευκορωσία ώστε να οδηγηθεί η χώρα στον εκδημοκρατισμό. πέραν από τη διατήρηση της σκληρής γραμμής της ευρωπαϊκής ένωσης για το υπάρχον καθεστώς και τη μη συμμετοχή της αντιπολίτευσης στην πολιτική σκηνή και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών η ένωση προσπαθεί να δεσμεύσει το σύνολο της κοινωνίας της λευκορωσίας για την επίτευξη του οράματος για τη δημιουργία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής χώρας. πρέπει όμως παράλληλα να διατυπωθεί σαφής πολιτικός στόχος για την εμπλοκή της ένωσης στη λευκορωσία με μια πιο συντονισμένη και προσεγμένη προσέγγιση ειδικά τώρα καθώς αντιμετωπίζει έντονα δημοκρατικά ελλείμματα. η περιφρόνηση των δημοκρατικών αξιών και του κράτους δικαίου όπως επίσης και η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η φυλάκιση πολιτικών της αντιπολίτευσης που παρατηρούνται σήμερα στη χώρα είναι καταδικαστέα και χρήζει ιδιαίτερη μεταχείρισης από την ένωση. Ευχαριστώ πολύ. λόγο κύριο Στάθνη 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην τελευταία συνάντηση με την αντιπολίτευση ε, θυμηθήκαμε πώς έχουν τα πράγματα εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ελευθερία στα δικαιώματα ε, δεν είναι σαν αυτά που έχουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν άλλη κατάσταση εκεί, δηλαδή ε, καταστολές παντός είδους, φυλακίσεις και κόσμους, πολίτες που ζουν διαρκώς υπό το κράτος του φόβου. Ο Λουκασέγκο ε, πηγαίνει, κάνει το γύρο του κόσμου, έχει περάσει από ψηφίσματα της Γερουσίας, ε, ψηφίσματα του Κοινοβουλίου. Ε, τον Ιανουάριο ο Ομπάμα κάλεσε στην, έτσι ώστε να υπάρξει πράξη και νόμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Λευκορωσία. Όλα αυτά τα Όλες αυτές οι νομοθετικές πράξεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να προωθηθεί η καταστροφή καταστολή ε, για ε, τον πολιτών. Ε, θα πρέπει και η Διεθνής Επιτροπή η Επιτροπή του Χόκκι Επιπαγού να πάρει την απόφαση να αλλάξει την έδρα των, του πρωταθλήματος στην επόμενη συνεδρίαση ε, στο ε, Ελσίνκι ελπίζω ότι θα συμφωνήσει και η Ομοσπονδία του Χόκκι Επιπάγου να αντιμετωπίσει την, ε, το νόμιμο αίτημα των δημοκρατών του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κρετού. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η επιδείνωση της καταστάσεως στην ε, Λευκορωσία ε, ολοκληρώθηκε κατά κάποιο τρόπο με τη μετάκληση των πρεσβευτών από το Μίνσκ. Ε, θα πρέπει όμως να ενθαρρυνθούμε να βρούμε μία λύση στην κατάσταση αυτή. Πρέπει να ζητήσουμε από την κυβέρνηση του Μίνσκ να σεβαστεί τα δικαιώματα των πολιτών και επομένως να αποκαταστήσει την την ε, ε, δημοκρατία. Θα πρέπει να ζητήσουμε να σταματήσει κάθε καταστολή και κάθε δίωξη ε, κατά των αντιπολιτευμένων, αντιπολιτευομένων και βεβαίως να ενστερνιστεί ε, η Λευκορωσία τις δημοκρατικές αρχές ε, που διέπουν την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γεγονός ότι οι πολίτες της Λευκορωσίας υποφέρουν από αυτή την κατάσταση καθώς επίσης και από την οικονομική ύφεση άνευ προηγουμένου. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους ομιλητές που έχουν ζητήσει το λόγο μέσω του Catch the Eye. Κυρία Εσάη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η αντιπολίτευση στη Λευκορωσία υφίσταται αφόρητη πίεση από τον πρόεδρο Λουκασένκο. Πολλοί ακτιβιστές και μέλη της αντιπολίτευσης δεν δικαιούνται να ταξιδεύσουν στην Αλλοδαπή, έχουν κατασχεθεί οι υπολογιστές τους, έχουν συλληφθεί οι ηγέτες της αντιπολίτευσης και μάθαμε προσφάτως ότι ε, μία οργάνωση δεν μπόρεσε να εγγραφεί στο Μητρό. Ζητήσαμε επιτακτικά την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Συμφωνώ με το αίτημα των κυρίων Αγιούλαντ και Στάσνη ότι θα πρέπει δηλαδή να ζητήσουμε ε, από την Διεθνή Ομοσπονδία Χόκκι Επιπάγου να ανακαλέσει τη διοργάνωση ε, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Χόκκι Επιπάγου από τη Λευκορωσία και την, να την αναθέσει σε άλλη χώρα. Αυτό δεν αφορά μποϊκοτάρισμα αθλητισμού. Θα πρέπει να γίνει αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά όχι σε μια χώρα ε, σαν τη Λευκορωσία και κυρίως όχι για να εξυπηρετήσει το κύρος και την έγκλη του Λουκασένκο. Η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι σχέσεις μας με τη Λευκορωσία φέρνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια παράδοξη και δύσκολη θέση. Είχαμε μεγάλες ε, εντάσεις διπλωματικές με πολύ γειτονική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η κατάσταση βέβαια θα αλλάξει όταν το καθεστώς του Λουκασέγκο σταματήσει να εφαρμόζει κατασταλτική πολιτική καταπίεση κατά των μελών της αντιπολίτευσης και κατά των πολιτών της Λευκορωσίας. Γιατί με την τακτική αυτή μόνο απομονώνει τη χώρα του οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα αναφέρουν στην έκθεσή τους ότι η Λευκορωσία περιλαμβάνεται στον κατάλογο χωρών που είναι εχθροί του ίντερνετ. Υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί στη χρήση του διαδικτύου στη Λευκορωσία. Και μάλιστα ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απέρριψε το αίτημα της Λευκορωσίας για δανεισμό. Φυσικά η τακτική αυτή του Λουκασέγκο ε, έχει ως πρώτο θύμα το πληθυσμό της Λευκορωσίας. Ελπίζω να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες ε, προς τον πληθυσμό της ε, Λευκορωσίας και να εξομαλυθούν το συντομότερο δυνατό οι σχέσεις μας με τη χώρα αυτή. Ο κύριος Λίζεκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Για πολλά χρόνια γίναμε όλοι μάρτυρες πολύ περίεργων σκηνών και του παιχνιδιού της γάτας και του ποντικού μεταξύ του ε, Λουκασέγκο που μια έκανε χαρούλες προς τη Δύση και μια προς την ε, Μόσχα ενώ ταυτόχρονα εφάρμοζε βίαιη καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης ε, των δημοσιογράφων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και μάλιστα το έκανε αυτό ασκαρδαμικτή. Ε, είχαμε και τη μετάκληση, ε, την κοινή απόφαση για μετάκληση των πρεσβευτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πρώτο σύμβολο μια ενιαία κοινή αντίδραση Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο των θεσμικών οργάνων, αλλά και των χωρών μελών. Και ήθε και στο μέλλον ε, να, δρούμε με την ίδια συνέπεια και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, δηλαδή και τα κράτη-μέλη απέναντι στο καθεστώ του Αλεξάνδρου Λουκασέγκο. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ε, Χόκκι Επιπάγου. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει ε, στο... Ε, στη Λευκορωσία δεν θα πρέπει να παίζουμε το παιχνίδι του Λουκασέκο και να του δίνουμε ευκαιρίε προβολή. Ο κύριο Νικολά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε στη διάσκεψη κορυφή Ανατολική εταιρική σχέση είχε αναλάβει την δέσμευση η ε, Λευκορωσία ότι θα σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θυμίζω ότι είναι μια χώρα γειτονική προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τόσο απομακρυσμένη όσον αφορά ε, τι αξίε. Πιστεύω ότι οι κυρώσει ε, θα πρέπει να εφαρμοστούν και στα πλαίσια τη Ανατολική εταιρική σχέση. Θα πρέπει να το συζητήσουμε με τα μέλη τη εταιρική σχέση, κυρίω δε με τι όμορε χώρε, έτσι ώστε να πιέσω με την κυβέρνηση του Μίνσκ για να αλλάξει στάση εάν ε, κάποιος ε, ε, σαν τον Λουκασέγκο αλλάξει δεν είναι σίγουρο. Εγώ γνωρίζοντας την προσωπικότητα του ανθρώπου έχω ισχυρές αμφιβολίες όσον αφορά το ενδεχόμενο αλλαγής της συμπεριφοράς του. Θα μπορούσαμε ίσως να συνεργαστούμε και με τη Ρωσία κατά την έννοια αυτή έτσι ώστε να δώσουμε και στην Ρωσία την ευκαιρία να δείξει την προσήλωσή της προς τις οικουμενικές αξίες. Ίσως η Ρωσία ουσία θα μπορούσε να στηρίξει ε, και να υπογράψει και τα ε, έγγραφα, τα σχετικά έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο έχει τώρα ο Επίτροπος κ. Πίκμπολς. Ε, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, Εξ ονόματος της ε, είπα της εκπροσώπου Άστον θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείξατε και τη δέσμευση που πάντα δείχνετε όσον αφορά τις σχέσεις με την Λευκορωσία. Ε, θέλουμε να εξακολουθήσουμε να βοηθούμε τη χώρα και τους πολίτες της. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ε, βοηθάει οικονομικά και πολιτικά την κοινωνία των πολλατών πολιτών καθώς επίσης ε, και την διασφάλιση των βασικών αρχών της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Επίσης ε, θα δοθεί η απαραίτητη οικονομική και λυπή στήριξη ε, προς τα θύματα αυτής της καταστολής. Στην κατάσταση που βρίσκονται μόνο από τη διεθνή βοήθεια μπορούν να περιμένουν κάτι. Επίσης θα πρέπει να ανοίξουμε ανοιχτές τις προοπτικές για τη χώρα. Ε, ε, περιοριστικά ε, μέτρα που τα οποία θα ληφθούν πρέπει και θα είναι στοχευμένα έτσι ώστε η πίεση να αφορά μονάχα την κυβέρνηση της Λευκορωσίας. Καθόλου δεν είναι στόχος μας να πλήξουμε τον, τους πολίτες της Λευκορωσίας. Προσωπικά πιστεύω και αυτό κατέστησα σαφές και από τη συζήτηση ότι το πιστεύουν όλοι δηλαδή και ορθώς ότι το μέλλον της Λευκορωσίας βρίσκεται στα χέρια των πολιτών της Λευκορωσίας. Ε, θα πρέπει να δράξουν την ευκαιρία έτσι ώστε να ε, ε, πάρουν πραγματικά τις απαραίτητες αποφάσεις και κατά αυτήν την έννοια βεβαίως όλες οι, συζητη... όλες οι αποφάσεις οι οποίες πρόκειται να ληφθούν θα συζητηθούν και βεβαίως πρέπει να πω ότι χαίρομαι που οι προτάσεις και τις υπά στηρίζονται και από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε έξι προτάσεις ψηφίσματος. Ε, ολοκληρώνεται τώρα η συζήτηση και επί των ψηφισμάτων θα λάβει χώρα η ψηφοφορία αύριο στις 12 το μεσημέρι. Έχουμε τώρα μία ανακοίνωση από τις ομάδες ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών